με θέμα ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνω το λόγο πρώτα στους ε, συντάκτες. Ε, ο κύριος Μάλκομ Χάρμπορ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Well, Mr. President, it gives me very great pleasure to present this. Χαίρομαι που η πολιτική μου ομάδα ηγείται αυτής της πρωτοβουλίας. Πρώτοι εμείς καταθέσαμε τη συγκεκριμένη πρόταση γιατί αυτό δείχνει πόσο σημασία δίνουμε στις αναπτυξιακές πολιτικές, σε αυτά τα μέσα τα οποία θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης στον τομέα της πραγματικής οικονομίας, χωρίς τεράστιες ροές επενδύσεων που έχουν ήδη κουράσει τους ταλαιπωρημένους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής θα πρέπει να δούμε τι ευκαιρίες υπάρχουν στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά Χαίρομαι που η ερώτηση του κυρίου Κρόιτσμαν ασχολείται με το ίδιο θέμα γιατί αυτό δείχνει ότι σκεφτόμαστε το ίδιο. Μιλάμε για μη εξερευνημένες δυνατότητες. Να υπάρξει εκκίνηση στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να υπάρξει απογείωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ιστορία δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιστορικά δημιουργούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης τα τελευταία δέκα χρόνια από οποιαδήποτε άλλη από οποιοδήποτε άλλο τομέα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν τις επιχειρήσεις αυτές να απογειωθούν σε όλες τις χώρες και να εκινεί η διαδικασία με αποτελεσματικό τρόπο. Ε, πολλές φορές είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν και τα υπάρχοντα μέσα. Τώρα για την ψηφιακή ε, εσωτερική αγορά, ενιαία μάλλον αγορά, κάθε εβδομάδα παίρνω μία έκθεση η οποία δείχνει τη σημασία των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές και το πόσο αυτό δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ την κυρία Ρέντινγκ για τον ρόλο τον οποίο έπαιξε όταν ήταν επίτροπος για τις τηλεπικοινωνίες απαιτείται να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να τονίσουμε, να ενισχύσουμε αυτές τις επενδύσεις, να μπουν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις στο διαδίκτυο. Οι τελευταίες εκθέσεις δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια στον κόσμο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν συνάδελφοι, έχουμε ευκαιρίες, έχουμε τα μέσα, γιατί δεν πιέζουμε τις κυβερνήσεις με τη στήριξη της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά και να δημιουργήσει αυτές τις νέες θέσεις απασχόλησης. Thank you. Ε, ευχαριστώ συνάδελφε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τόμας Χέντελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και χρόνια διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αλόγιστη πολιτική εξοικονομήσεων σε βάρος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία έχει οδηγήσει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σημαντική οικονομική ύφεση και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι παραγνωρίζεται το γεγονός ότι είναι σημαντική η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και χωρίς οικονομική δραστηριότητα δεν μπορεί να υπάρξει καμία ίσπραξη φόρων και καμία κοινωνική ε, πρόοδος. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να προέλθει μόνο από τη λιτότητα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη δεν είναι μία μονάχα φυσαλίδα, μία πομφόλιγα, αλλά είναι ένα σύνολο από συγκεκριμένα και στοχευμένα προγράμματα. Το τελευταίο πρόγραμμα της Κομισιόν για το 2013, εγώ είδα πάρα πολύ ωραίες ε, φράσεις ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει με την ε, κοινωνική οικονομία της αγοράς, τις προκλήσεις της ε, εποχής και μπορεί πάντα να μπορεί να είναι στην αιχμή του δόρατος της νέας Βιομηχανική επανάστασης. Μα αγαπητοί μου συνάδελφοι, αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο ότι θα υπάρξει περαιτέρω αποδόμηση του κοινωνικού κράτους για μεγαλύτερη κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε προς την ίδια κατεύθυνση με τον ίδιο ρυθμό να, κατα... <clears throat> να καταστρέφουμε τον ιστό της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας οι οποίες θα μπορούν να εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό είναι απαραίτητο για το μέλλον των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε από μια Ευρώπη η οποία βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στον ανταγωνισμό προς μια Ευρώπη η οποία βασίζεται και στην αλληλεγγύη. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο να κοιτάζουμε τους ισολογισμούς, θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία θα είναι και δίγεια σε φορολογικό επίπεδο και που θα κάνει και τους πλούσιους στην Ευρώπη να επομιστούν ένα τμήμα του συνολικού φορολογικού βάρους. Αυτό σημαίνει επίση μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, η οποία δημιουργεί θετικέ θέσει εργασία, παραδείγματο χάρη με την αλλαγή στον ενεργειακό τομέα και την προστασία της, του, από την κλιματική αλλαγή. Η Γερμανική Ένωση Συνδικάτων έχει ζητήσει, έχει παρουσιάσει μάλλον ένα νέο πρόγραμμα Marshall, ένα σχέδιο Marshall για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει αυτήν την ε, διαδικασία. Το να είμαστε στην αιχμή του δόρατος της βιομηχανικής επανάστασης αυτό έχει νόημα μόνο όταν δίνει στους πολίτες ένα καλύτερο μέλλον και όχι μονάχα όταν ενισχύει τα θυλάκια των πλουσίων. Γι' αυτό εμείς πρέπει ως Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε κυρία για λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οικονομική κατάσταση της Ένωσης και οι προοπτικές ε, της ΟΝΕ για το 2013 είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει με αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Δεν θα πρέπει η ιδεολογία να επιβάλλει λιτότητα ανελαίτη. Από το 2008 προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την κρίση και από το 2010 είχαμε τι πολύ αυστηρέ πολιτικέ τη λεγόμενη δημοσιονομική εξηγήση που εφαρμόστηκαν με πολύ βίο τρόπο στι πιο εύθραυστε και βάλωτε οικονομίε. Σήμερα έχουμε ήδη κάποια αποτελέσματα. Οι προβλέψει πέρυσι έλεγαν ότι το 2011 ε, η Ελλάδα θα αναπτυχθεί κατά 0,7% αλλά έπεσε σε ύφεση 6,9. Ε, η Πορτογαλία που τήρησε ευλαβικά τις συστάσεις της Τρόικας αναμενόμενη ανάπτυξη για το 2011 ήταν 0,7%. Τελικά κατέληξε και κίνησε ε, ύφεση μείον 1,7%. Όπως είχαμε προβλέψει πριν από δύο χρόνια, οι πολιτικές λιτότητας, οι συγχρονισμένες αυτές πολιτικές που καλύπτουν χώρες που έχουν... που έχουν πλεονάσματα και άλλες που έχουν ελλείμματα, δεν ε, οδηγεί σε δημοσιονομική εξυγίαση, αλλά δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο σιγά σιγά ακόμη και πιο ισχυρέ οικονομίε αρχίζουν και λυγίζουν. Και ενώ περιμέναμε φέτο να αναπτυχθούμε κατά 0,5% θα, θα καταλήξουμε να έχουμε απώλεια του πλούτου 0,04% και ύφεση. Και 25 εκατομμύρια πολίτες είναι χωρίς απασχόληση, οι νέοι απελπισμένοι και οι πολίτες αρχίζουν να χάνουν τις ελπίδες τους για το κατά πόσο πιάνουν τόπο αυτές οι θυσίες που έκαναν. Και θα πρέπει να αλλάξουμε τη ρητορική μας ότι μερικοί είναι αμαρτωλοί και άλλοι είναι ενάρετοι. Θα πρέπει να δούμε τη λύπη από το αρχιτεκτόνημα τη ΟΝΕ. Προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά και τις αδυναμίες, αλλά από τις παρατηρήσει παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να αντλήσουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Η συνταγή της δημοσιονομικής εξυγίασης αν δεν αναθεωρηθεί ε, ριζικά δεν θα έχει καλά αποτελέσματα και θα πρέπει να παραταθούν τα χρονοδιαγράμματα της δημοσιονομικής εξηγίασης. Θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή η δημοσιονομική εξυγίαση, αλλά με ρεαλιστικό τρόπο, με ε, τόκους που θα είναι όσο πιο μικρή γίνεται και χωρίς ε, ε, επιβράβευση εκείνων που χρηματοδοτούν τις χώρες. Σε ό,τι αφορά την ε, οικονομία, σε περίπτωση που μπαίνει σε ύφεση θα πρέπει να περιορίζεται η λιτότητα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Σήμερα αναγνωρίζουμε ότι η τα δάνεια, τα κεφάλαια δεν φτάνουν στην πραγματική οικονομία. Και η ευρωπαϊκή πολιτική δεν έχει μια γνήσια βιομηχανική πολιτική. Ούτε έχουμε μια πραγματική εξωτερική εμπορική πολιτική που θα προσαρμόζεται στο παγκοσμιοποιημένο μα περιβάλλον. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με σταθμισμένο και ισορροπημένο τρόπο και ορθολογικό θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση. Να μην ξεγελαστούμε από ομιλίες ούτε από πολιτικές που στόχο έχουν να, δικαιολογήσουν τα κακό κείμενα. Η κατάσταση είναι υπερβολικά σοβαρή. Έχουμε τεράστια ανεργία, απώλεια προοπτικών. Οπωσδήποτε λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις συνταγές που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Κυρία είχε είχε Κρόιτσμαν, Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Κρότσμα για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε Ρέντινγκ, συμφωνώ και με τον, τους προλαλήσαντες ότι είναι πολύ σημαντική ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θα πρέπει όμω να εξασφαλίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα προσθέσουμε πρόσθετη γραφειοκρατία. Αντίθετα θα την μειώσουμε γιατί επηρεάζει αρνητικά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Χρειαζόμαστε ένα σύμφωνο ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό όμω προποθέτει ότι θα έχει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα προ αυτό και αγαπητέ συνάδελφε κύριε Χέντελ, δεν χρειαζόμαστε πάλι των τάξεων. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ευκαμπτοποίηση της ε, αγοράς εργασίας γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μια ανεργία 50% στην ε, Ελλάδα και στην Ισπανία, 30% στην Ιταλία και τη Γαλλία ανεργία των νέων. Είναι απαραίτητο λοιπόν εμείς να μπορέσουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στους νέους να εργαστούν, να δώσουμε να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον χώρο εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να περιστήλουμε και την ανεργία μέσα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από τις ρητορικέ εκρήξεις για την πάλη των τάξεων και θα παίξει και πιο θετικό ρόλο μέσα στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις σε σχέδια υποδομών. Πολύ σωστά αναφέρθηκαν οι μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και αυτοί οι τομείς θα πρέπει να τύχουν και ιδιωτική πρωτοβουλίας και συμβολής να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα απαραίτητα πρέπει ώστε να είναι πράγματι ελκυστικές αυτές οι επενδύσεις και να υπάρξει και η απαραίτητη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το σύμφωνο αυτό ανάπτυξης θα είναι πραγματικά μια ευκαιρία για όλους αν αφήσουμε κατά μέρο όλα τα αρνητικά στοιχεία της ενιαίας αγοράς και όταν μπορέσουμε, όπως ζητούμε συνέχεια στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, να περατώσουμε την δημιουργία της εσωτερικής αγοράς και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και νέες ευκαιρίες απασχόλησης για τους πολίτες Ευρώπης. Ευχαριστώ. Κύριε, Θα δεχτείτε ένα ερώτημα, μια μπλε κάρτα από τον κύριο Χέντελ. Δεν κατάλαβα τι εννοούσατε κύριε Κρόισμαν όταν μιλήσατε για πάλι των τάξεων σε σχέση με τη δική μου παρέμβαση. Αν θεωρείτε πάλι των τάξεων το ότι όλο περισσότερο κερδίζει ο ιδιωτικός τομέας ενώ ο δημόσιος τομέας και η απασχόληση χάνει, τότε δεν έχετε καταλάβει καθόλου αυτό το οποίο εννοούσα. Κύριε Χέντελ, δεν έχει νόημα να αναφέρετε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα. Οι θέσει εργασία δημιουργούνται από την οικονομία. Όταν υπάρχουν ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά, τότε μπορούν να δημιουργηθούν και μόνο θέσει εργασία από τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Έχουμε 25 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και εισάριθμους ανέργους. Αν κάθε μικρομεσαία επιχείρηση μπορούσε να δημιουργήσει μια θέση εργασίας, θα είχαμε ξεπεράσει το πρόβλημα. Σας λέω πάντα, αν είχαμε και μία αντιμετώπιση στη Γερμανία που να είναι σαν αυτή που έχουμε με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχαμε λύσει πάρα πολλά περισσότερα προβλήματα. Αυτά που λέτε εσείς θα οδηγούν σε λύσεις. την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θυμηθείτε ότι πρόκειται για τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και μέσω πρόθεσμα και βαχυπρόθεσμα, ε, διατηρώντας πάντα τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί τώρα στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη. Τα στοιχεία είναι πλέον διαθέσιμα. Θα πρέπει απλά να προωθήσουμε τα μέτρα τα οποία έχουν επεταθεί, όπως το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, οι συμφωνίες, τα Σύμφωνα για την Ενία, Αγορά 1 και 2, όπως επίσης και οι προτεραιότητες ε, για την έρευνα ανάπτυξης αιτήσια το 2013. Ξέρουμε ότι τα μέτρα αυτά είναι επιμέρους συγκεκριμένα μέτρα. Γνωρίζουμε ότι το θέμα, το πραγματικό, το ουσιαστικό της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εφημερίας θα αντιμετωπιστεί μόνο αντιμετωπίζοντας τα διαφορετικά προβλήματα των οικονομιών μας. Σταθεροποίηση της ζώνης ευρώ, ίσως το πιο επίγον θέμα στην παρούσα συγκυρία, αντιμετώπιση όλων των απαραίτητων μέτρων για να εμπνεύσουμε πλέον εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία, διότι αν δεν υπάρξει αίσθηση εμπιστοσύνης δεν θα υπάρξουν επενδύσεις και αν δεν υπάρξουν επενδύσεις δεν θα υπάρξουν δυνατότητες για ανάπτυξη και φυσικά η ανάπτυξη είναι η απάντηση. Αυτό το οποίο λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με αποφασιστικότητα και στα πλαίσια της ανάληψης ευθυνών και στα πλαίσια της εφαρμογής της αλληλεγγύης απαιτούνται μεταρρυθμίσεις για να ε, προχωρήσουμε στην αηφόρο ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και γι' αυτό η Επιτροπή στα πλαίσια της ε, μελέτης της, της έρευνάς της για το 2013 υπογραμμίζει τις εξής πέντε προτεραιότητες. Πρώτον, διαφοροποιημένη ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Δεύτερον, αποκατάσταση της δυνατότητας δανειοδότησης της οικονομίας. Τρίτον, προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας για το σήμερα ή για τον επόμενο χρόνο με την αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κατάστασης. Και τέλος, εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Στον τελευταίο τομέα, σαν παράδειγμα, πολλά μπορεί να γίνουν στον τομέα της ψηφικοποίησης της δημόσιας διοίκησης, των δημοσίων προμηθειών, της βελτίωσης της ανεξαρτησίας των δικαστικών συστημάτων καθιστώντας ε, ε, έτσι ικανά τις δικαστικές διαδικασίες καθιστώντας τις ικανές να προωθήσουν την προσπάθεια αυτή. Έτσι θα μπορέσουμε να ωφεληθούμε από τα επιτεύγματά μας και ακριβώς επειδή τα προγράμματα αυτά είναι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, απαιτούνται και βραχυπρόθεσμοι πρωτοβουλίες για να υπάρξουν άμεσες επενδύσεις. Και εδώ ε, φυσικά παίζει ρόλο ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι ένα μέσο για επενδύσεις, είναι ένα μέσο για επενδύσεις στο σύνολο της Ευρώπης. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για την ανάγκη για ανάπτυξη χωρίς να αναγνωρίσουμε την κρίσιμη ανάγκη για στοχευμένε επενδύσεις ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το σημαντικότερο μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Εάν εμείς θέλουμε πράγματι να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να υπάρξουν σωστοί ε, προϋπολογισμοί που θα διευκολύνουν ε, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Γι' αυτό απαιτείται άμεσα συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τους ευρωπαϊκούς μοχλούς ανάπτυξης. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα εργασίας για το 2013 αναφέρεται σε συγκεκριμένες σημαντικές πρωτοβουλίες που ήδη έχουν γίνει και κάνει επίσης και κάποιες νέες συμπληρωματικές. Θα, συνεχίζω, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα επικοδομητικά με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έτσι ώστε οι προτάσεις αυτές να γίνουν δεκτές και νομίζω ότι αυτό είναι βασική προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, έχει εκφράσει τις θέσεις και για τους λεγόμενους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Απαιτείται να υπάρξει δηλαδή μια έξυπνη μορφή συνδυασμού των μέτρων για τη δημοσιονομική εξυγίανση, να διευκολύνουμε τις οικονομίες οι οποίες έχουν χάσει την πρόσβασή τους στις διεθνείς χρηματαγορές. Δεν υπάρχει δυνατότητα εδώ αναβολής της λήψης αυτών των μέτρων. Για τις χώρες οι οποίες έχουν περισσότερη δημοσιονομικά περιθώρια, οι αυτόματοι σταθεροποιητές καλούνται να παίξουν το σημαντικό τους ρόλο Σχετικά με τα υπάρχοντα πλεονάσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σε αυτή τη φάση μια οριζόντια ανάλυση των πολιτικών συνεπειών τέτοιου είδους πλεονασμάτων μικρών και μεγάλων και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής αναμένονται ε, τους πρώτους μήνες ε, του 2013 και θα στηρίξουν τεκπηριώνοντας και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τώρα, για την αύξηση του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι διοικητές της τράπεζας αυτής θα εγκρίνουν επίσημα την αύξηση κατά ένα δις τις επόμενες εβδομάδες. Και το πρόγραμμα δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τα επόμενα τρία χρόνια θα αντικατοπτρίζει τις αυξημένες δανειοδοτικές ικανότητες της συγκεκριμένη τράπεζας. Είναι σαφές ότι είμαστε μια οικονομική ένωση, έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα, έχουμε την δυνατότητα να ε, εμβαθύνουμε την ενιαία μας αγορά αλλά στόχος μας πάντα παραμένει ένας στόχος πολιτικός και κοινωνικός. Οι πολίτες. Συναντιέται, ξέρετε, σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους δρόμους για μια πιο γνήσια και ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση Καλούμεθα λοιπόν να ακούσουμε και τις απόψεις του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια Ευρώπη σταθερή, ισχυρή, αλληλέγγυα και δημιουργική στον τομέα της απασχόλησης. Ευχαριστώ, πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν. Ε, ακολουθούν οι ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Για το ΕΛΚ έχει το λόγο ο κύριος Ανδρέας Σβάβ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για την ανάπτυξη στην Ευρώπη έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση με αυτά τα οποία μόλις ανέφερε η κυρία Ρέντινγκ από ότι από αυτά που ακούσαμε από τους συναδέλφους. Η Ευρώπη και η ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, πλήττεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην εσωτερική αγορά και πολύ λιγότερο οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγους κανονισμούς. Για μένα η μεταρρύθμιση και η ανάπτυξη μπορούν να προέλθουν όταν έχουμε ένα ενιαίο χώρο σε όλη την Ευρώπη, ο οποίος όμως είναι λειτουργικός. Αυτό το οποίο βλέπουμε αντίθετα είναι ότι χώρες όπως η η Ελλάδα και η Πορτογαλία, για να γυρίσω στην κυρία Φερέιρα, έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι πραγματικά πρωτοποριακού χαρακτήρα. Ο ΩΣΑ έχει κατατάξει χώρες όπως είναι η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα σε χώρες που είναι πρωτοποριακές σε ό,τι αφορά την ταχύτητα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι επαρκής αυτή η διαδικασία μεταρρυθμίσεων για να οδηγήσει στην ε, ε, ανάπτυξη εάν δεν υπάρχει και η σωστή εφαρμογή τους. Και γι' αυτό τονίζω αυτά τα οποία είπε η κυρία Ρέντι. Χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή, καλύτερη λειτουργία αυτών των κανόνων και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια καλύτερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, μια καλύτερη διακυβέρνηση της οικονομικής μεταρρύθμισης. Δεύτερον, πιστεύω ότι η ανάπτυξη μπορεί να προκύψει μονάχα όταν έχουν εμπιστοσύνη και οι πολίτες για την οικονομική ανάπτυξη και είναι σίγουροι ότι τα μέτρα τα οποία εμεί έχουμε αναλάβει και τα οποία αρχίζουν να αποδίδουν ε, αποτελέσματα στην Ευρώπη, παραδείγματο χάρη βλέπουμε στην Ελλάδα ότι επανέρχεται στι χρηματαγορέ, ότι αυτά τα μέτρα θα αποδώσουν καρπού. Εάν δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη των ανθρώπων δεν θα ευδοκιμήσουν. Και δεν πρέπει εμείς να διστάζουμε για το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα και να αλλάζουμε κατεύθυνση. Όχι, αν προχωρήσουμε με σταθερό βήμα και εφαρμόσουμε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τότε η Ευρώπη θα ξαναβρει τον δρόμο της. Α, η κυρία Φερέιρα θέλει να κάνει χρήση μπλε κάρτας. Ναι, ναι. κυρία Ευχαριστώ κύριε Σουάμπ. Θα ήθελα να σας θέσω το εξή ερώτημα. Κατανοείτε ότι τα πλεονάσματα της Γερμανίας προκύπτουν από το γεγονός ότι το νόμισμα της Γερμανίας δεν έχει ανατιμηθεί γιατί είναι το κοινό νόμισμα όλης της Ευρώπης ενώ άλλες χώρες είναι χώρες που θα έπρεπε να είχε υποτιμηθεί το νόμισμά τους. Κατανοείτε ότι η Γερμανία έχει ε, χρηματοδοτήσει τι εξαγωγέ τη μόνο με την χρέωση, την υπερχρέωση των χωρών της περιφέρειας. Κύριε Σβάμπ. Χωρί μικρόφωνο κύριε Σφάμπ. Κυρία Φερέρ, σας ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα. Εγώ δεν διαφυσβήτησα ποτέ και ούτε οι Γερμανοί θα το κάνουν ότι η ενιαία αγορά και η συνεργασία στην Ευρώπη έχουν σταθεί ιδιαίτερα θετικές για την Γερμανία. Και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι για μια αλληλεγγύη με τις άλλες χώρες στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι το πρώτο βήμα είναι η μεταρρύθμιση και το δεύτερο βήμα θα πρέπει να, εξασφαλίσουμε μια ενότητα στην Ευρώπη και μια αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε για με μέτρα τα οποία θα ανατρέψουν και πάλι την οικονομική πρόοδο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει και φυσικά θα πρέπει να συνοδεύεται αυτός ο δρόμος και από αλληλεγγύη. Ε, για την ε, ομάδα S&D το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Αλεχάνδρο Θέρκας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρέντε, κύριε Επίτροπε, ε, μιλήσατε στο τέλος της ομιλίας σας για μια Ευρώπη που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Το πρόβλημα όμως, κύριε Επίτροπε, είναι ότι στην Ευρώπη χάθηκαν 2 ε, εκατομμύρια θέσεις εργασίας το τελευταίο, το τελευταίο χρόνο και αυτά τα 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ήδη ε, επηρεάζουν τους μακροχρόνια ανέργους, τους ε, νέους που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Έχουμε ένα πρόβλημα που διαιωνίζεται, είναι πια χρόνιο, διαρθρωτικό. Έχετε αυτή την ανησυχία, αλλά εμεί έχουμε μια επιπλέον ανησυχία. Ε, Δεδομένη αυτή τη πραγματικότητα, εσεί επιμένετε στα προτινόμενα μέτρα. Μα μέχρι πότε, κυρία Ρέντινγκ, μέχρι πότε θα συνεχίζουμε να εκτελούμε, όπω λέμε στα Ισπανικά, γιατί αυτό κάνετε ουσιαστικά. Εκτελείτε τι χώρε του Νότου. εκτελείτε μια ολόκληρη γενιά με τι πολιτικέ τη λιτότητα που δεν συνοδεύονται από αναπτυξιακέ πολιτικέ. Μέχρι πότε λοιπόν θα περιμένουμε και θα συσσωρεύουμε στοιχεία τραγωδιών οικονομικών και κοινωνικών ε, για να αλλάξουμε πόρια. Είναι μια κατακραυγή που ακούμε από το λαό που δυστυχώς προσκρούει σε κοφά ότα στο Συμβούλιο που έχουν ε, ορθώσει τύχη και δεν ακούν τίποτα. Πότε θα ε, εφαρμόσετε κάποιες αντισυγκυριακές, αντικυκλικές πολιτικές. Αν δεν κάνετε κάτι τέτοιο θα συνεχίσετε να επιτείνετε την ανεργία και την εξαθλίωση. Πώς θα προσπα... προστατεύσουμε ένα κοινοτικό προπολογισμό δεν έχει επενδύσει και αν περικόπτονται συνέχεια τα κονδύλια του και συρρυκνώνεται. Πώ θα έχουμε εμπιστοσύνη μια πολιτική που μα οδηγεί στην καταστροφή. Όπω είπε η κυρία Φεραίρα, ε, δεν ε, ζητάτε ε, να συνεχιστεί να αυξάνεται η ζήτηση όχι μόνο στις χώρες που έχουν πλεόνασμα αλλά και στις χώρες που έχουν έλλειμμα που εκεί καταπνίγεται η ζήτηση. Καταστρέφεται η ζήτηση, καταστρέφεται η ζωή των ανθρώπων, καταστρέφονται οι επιχειρήσεις, χάνονται χιλιάδες ε, θέσεις απασχόλησης. Ζητήσατε ελαστικότητα, να μα εσείς πρώτα να την εφαρμόσετε εκεί και να μας δίνετε στοιχεία και να μην ενδίδετε σε ιδεολογικές προκαταλήψεις. Ευχαριστώ. Συνάδελφος κύριος Μάντερς για την ομάδα των για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εδώ και πολύ καιρό μιλάμε για ανάπτυξη στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι είναι η μαγική λέξη. Ανάπτυξη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τι γίνεται όμως με την εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών και των καταναλωτών στο μέλλον της ενιαίας αγοράς. Θα πρέπει να συντρέξουν κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους οι επιχειρηματίες και οι καταναλωτές και να δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο για να μπορούν και οι καταναλωτές αλλά και οι επιχειρήσεις ε, να κάνουν τον προγραμματισμό τους και να χαράζουν τη στρατηγική τους. Τέτοιες προϋποθέσεις θα πρέπει να διασφαλιστούν με την ευρωπαϊκή πολιτική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δυστυχώς, ε, πολλές ε, νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται ως προτάσεις που εμποδίζουν, παρεμποδίζουν την ανάπτυξη. Άλλωστε έχουμε και οδηγίες που εφαρμόζονται ε, γι' αυτό και δημιουργούνται τεράστιες διαφορές στην ενία αγορά. Θα προτιμούσα λοιπόν να έχουμε οδηγίες που θα είναι πιο αποτελεσματικές, που θα εφαρμόζονται πιο σωστά και ομοιόμορφα, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την ε, ενωσιακή νομοθεσία σε λίγη και καλή σε λειτουργικές νομοθετικές πρωτοβουλίες ε, που θα ευνοούν και τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές. Μιλήσαμε και για τις επιχορηγήσεις. Μα οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις είναι σαν υπνοτικό. Δεν δίνουν ενάυσματα για την καινοτομία. Είναι απλώς σαν παυσίπονο. Και μιλήσαμε για την καινοτομία. Με την καινοτομία θα δημιουργήσουμε εργασία. Ε, η το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος για ένα λεπτό. Iš tiesų taupimo priemonės įtraukė ekonomiką į pavojingą nuosmukį. Κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι η λιτότητα μας οδήγησε σε ένα πολύ επικίνδυνο καθοδικό σπιράλ. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά και μερικές φορές αρνητικά. Έχουμε μια κούρσα, έναν αγώνα δρόμου που προσπαθούμε απελπισμένα να αυξήσουμε το ΑΕΠ, έστω και ελάχιστα, αλλά τελικά έχουμε μια ελεύθερη πτώση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, να το κρατήσουμε σταθερό, αλλά δυστυχώς ε, η ύφεση επιτείνεται θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η λιτότητα δεν ε, μας έχει οδηγήσει πουθενά, δεν έχει βελτιώσει σε καμία περίπτωση την οικονομία μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Καταρχήν να ενισχύσουμε, να τονώσουμε την παραγωγή και την κατανάλωση, να επενδύσουμε στις, ε, στην εξοικονόμηση, αλλά να μην ε, επιβάλλουμε θυσίες στους συμπολίτε, απλώς να περικόψουμε τη γραφειοκρατία μας και επίσης να γίνει πιο αποτελεσματική η πολιτική μας με σωστές δαπάνες. Επόμενος ομιλητής, εξ ονόματο της ομάδος της Γκουε, είναι ο συνάδελφο κ. Νικόλαος Χουντή και έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ας μιλήσουμε λοιπόν για ανάπτυξη στην Ευρώπη, πράγμα που προκάλεσαν οι ερωτήσεις που κατατέθηκαν. Για ανάπτυξη ως απάντηση στην ύφεση. Σε μια ύφεση που είναι πρωτοφανών διαστάσεων σε όλη την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι εικόνε, κυρία Επίτροπε, που εμφανίζουν ιδιαίτερα ορισμένε χώρε του νότου με υψηλή ανεργία με παιδιά που υποσυντίζονται, με οικογένειε που χάνουν τα σπίτια του σα είναι γνωστέ. απάντηση βεβαίω είναι η ανάπτυξη αλλά οι πολιτικέ που ακολουθούνται ερμηνεύουν την κρίση με διαφορετικό τρόπο ενώ είναι κρίση των νεοφιλελεύθερων μοντέλων επιμένουν σε αναποτελεσματικέ πολιτικέ και αυτά που μα εξαγγείλατε με καλέ προθέσει κυρία ρέντινγκ ω αναπτυξιακέ πολιτικέ που βλέπει η κομισιόν είναι μια απλή ρητορική και είναι και αναποτελεσματική. με παράδειγμα την ελλάδα που χρησιμοποιήθηκε ως πειραματόζω εφαρμογής αυτών των πολιτικών διεξόδων από την κρίση η κατάσταση αυτή γενικεύτηκε η μία μετά την άλλη οι χώρες μπαίνουν σε μνημονιακές πολιτικές σε πολιτικές λιτότητας τα αποτελέσματα για όλη την ευρώπη είναι γνωστά δεν τα αναφέρω δείτε τα στοιχεία της eurostat. κυρία επίτροπε ακούστε τώρα τα οξύμορα και τα ε, αντιφατικά των πολιτικών που υποτίθεται ότι βοηθούν την ανάπτυξη. σημείο πρώτο σύμφωνα με το πολιετές δημοσιονομικό σύμφωνο για την ελλάδα αναφέρομαι και για άλλες χώρες προφανώς μια χώρα που έχει χάσει 25% λόγω της ύφεσης του αεπ που έχει 26% ανεργία περικόπτονται κατά το μισό τα έσπα. η κομισιόν επικαλείται ότι δεν το επιτρέπουν οι κανονισμοί να κάνει διαφορετικά όμως αυτούς τους κανονισμούς μπορούσατε να τους αλλάξετε πώ λοιπόν μπορεί να περιμένει μια αναπτυξιακή όθηση μια τέτοια χώρα και προφανώ και άλλε χώρε. σημείο δεύτερο αναφέρθηκε ο κύριο συνάδελφο λέει μεταρρυθμίσει που λαμβάνονται στι χώρε του νότου. τι εννοεί αυτό. η πολιτική τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη ανταγωνιστικότητα ε, πλήττουν ευθέω την ανάπτυξη. το παράδειγμα είναι πολύ συγκεκριμένο. στην ελλάδα παρά την εσωτερική υποτίμηση παρά την περικοπή των μισθών οι επιχειρήσει φεύγουν λόγω περιορισμένη ζήτηση και λόγω ευρωπαϊκή πολιτική που αυξάνει το ρίσκο. επομένω αυτέ οι πολιτικέ είναι αναποτελεσματικέ πρέπει να ακολουθούν διαφορετικέ πολιτικέ με αυτέ δεν θα πετύχουμε την ανάπτυξη. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χουντή. Ε, μεταβαίνουμε τώρα στου ε, άλλου εγγεγραμμένου ομιλητέ και δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Πάουλο Ρανζέλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να χαιρετήσω τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται από την Κομισιόν είτε σε φραστικό επίπεδο σε επίπεδο μέτρων για μια στρατηγική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χωρεί αμφιβολία για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα συνειδητοποιημένη σε σχέση με την ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη. Τα σχέδια που οι προτάσει που έχει υποβάλει κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, θα θέλω να υπενθυμίσω το εξή. Η στρατηγική αυτή η οποία έχει χαραχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια στρατηγική μέχρι το 2020 για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά οι χώρες του μνημονίου και άλλες χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι σε μεγάλη δυσκολία σε σχέση με τι οικονομίε του. Πρέπει να χαιρετήσουμε την προσπάθεια που γίνεται για την εξυγίανση των οικονομικών, αλλά χρειάζεται μια πρόσθετη βοήθεια για την ανάπτυξη. Δηλαδή, η στρατηγική ανάπτυξή μα θα πρέπει να είναι μια συνολική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και ιδιαίτερα μέτρα τα οποία είναι <clears throat> εστιασμένα στην ανάπτυξη των χωρών που βρίσκονται στη διαδικασία εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών του. Πέραν αυτών τα οποία ελέγχθηκαν εδώ, επομένω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτή η πραγματικότητα τη Ελλάδα τη Πορτογαλία, τη Ιρλανδία, χωρών όπως είναι η Κύπρος, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Ιταλία που χρειάζονται αυτή τη στιγμή μια πιο προσεκτική αντιμετώπιση των προβλημάτων τους σε σχέση με την ανάπτυξη, όχι με την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, αλλά ακριβώς με την ανάπτυξη. Και εδώ θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή τη στιγμή έχει γίνει αυτή η αύξηση κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και δεύτερον, αν κάποια από τα σχέδια θα τύχουν προτεραιότητες για τις χώρες, ιδίως της περιοχής που έχουν προβλήματα ύφεσης. Ραζέλ, επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Χουάνγκ Γκόγκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ρέντινγκ, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Επίτροπος Ρεν υποστήριξε σε δήλωση στον τύπο ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι ευεργετικές. Τα επιχείρημα αυτό το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στην ετήσια έκθεσή σας, μας εκπλήσει. Όπου εφαρμόζεται αυτή η πολιτική δεν, επέτρεξε, δεν επέτρεψε συγγνώμη, να επιτευχθούν οι στόχοι για τη μείωση των ελλημάτων. Η Ελλάδα μείωσε τα έξοδά της, μείωσε ε, τους ε, μισθούς έπρεπε να είναι τρομερά ανταγωνιστική και είναι η πλέον απελπισμένη κοινωνία της Ευρώπης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε επίσημα ότι ε, υποτίμησε την υφεσιακή επίπτωση των πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης που προτάθηκαν από την Τρόικα. Είπαν ότι οι πολλαπλασιαστές είναι μεγαλύτεροι από ό,τι πίστευαν. Αν φτάσει το 1,5 τότε θα έχουμε μία μείωση δαπανών κατά 10 που κάθε φορά θα συρρυκνώνει το ΑΕΠ κατά 15 δις. Σχετικά τώρα με τις επιπτώσεις στον τομέα της εμπιστοσύνης, προφανώς δεν έχουμε τίποτα το θετικό ακόμα. Είναι σαφές ότι η Γενική Διεύθυνση Έξιν είναι απόστολος των λεγόμενων ισοτιμιών του Ρικάρδο, όπως λέγονται στην οικονομική θεωρία κάτι το οποίο θα επιτρέψει υποτίθεται στις κοινωνίες αυτές να αυξήσουν την ε, ζήτηση και τις επενδύσεις τους. Όπου όμως έχουν μειωθεί οι δημόσιες επενδύσεις για να μειωθούν και οι φόροι, αυτό δεν έχει σε καμία περίπτωση επηρεάσει την αύξηση της ύφεση. Και τέτοιου είδους δημοσιονομικά μέτρα δεν επέτρεψαν τη μείωση των ελλημάτων. Το λάθος της Γενικής Διεύθυνσης ΕΞΥΜ προέρχεται από το ότι τα πρότυπα τα οποία χρησιμοποιεί αγνοούν την ύπαρξη των λεγόμενων πολλαπλασιαστών. Από επιστημονική ανεπάρκεια, από άγνοια ή από ιδεολειψία για νεοσυντηρητικές πολιτικές αρνείται η απο ιδεολειψια για νεο συντηρητικες πολιτικες Επιτροπή να αλλάξει τις ε, προοπτικές της όπως το έχει ήδη κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι επιλογές αυτές οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερε. και γι' αυτό η ετήσια έκθεση της Κομισιόν τον επόμενο χρόνο πρέπει να γίνει αντικείμενο κοινοβουλευτική έκθεσης, νομοθετικής έκθεσης. Η κυρία Χίρς έχει το λόγο για ένα λεπτό αλλά και 30 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε Ρέντινγκ. Ως ε, εκπρόσωπος της Κοινωνικής Επιτροπής θέλω να αναφερθώ στα θέματα της ανάπτυξης. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας στην Επιτροπή Απασχόλησης. Η πιο κοινωνική πολιτική που μπορεί να ασκηθεί είναι το να δώσουμε στους ανθρώπους θέσεις απασχόλησης. Αυτό το έχουμε τονίσει πάντα στην Επιτροπή Απασχόλησης. Είναι απαραίτητο να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και είναι οι επιχειρήσεις φυσικά οι οποίες θα δημιουργήσουν αυτέ τι θέσει απασχόληση και όλο ιδιαίτερω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει οι οποίε δημιουργούν τι θέσει απασχόληση. Είναι απαραίτητο να έχουμε κοινωνικά προγράμματα, αλλά αυτά μπορούν απλώ να γεφυρώσουν ένα χρονικό διάστημα. Εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα είναι η δημιουργία απασχόληση, και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε ευνοϊκότερε συνθήκε για τι επιχειρήσει και ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν και όλοι οι κανόνες και οι νομοθετικοί κανόνες στους οποίους έχουμε ήδη εγκρίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι ότι πάντα είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν περαιτέρω ρυθμίσεις και στις χώρες όπου λειτουργούν. Θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσουμε ότι επιτέλους θα βρούμε έναν τρόπο να εφαρμόσουμε πλήρως το σύνολο των κανόνων που οδηγούν στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και επομένως να δημιουργήσουν και ε, ανάπτυξη. Πιστεύω ότι σε πολλού τομεί, ιδίω στον τομέα των μέσων ενημέρωση, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να έχουμε περαιτέρω ανάπτυξη και απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χίρ. Ο κύριος Σιμάνσκι. For one minute. Κύριε Πρόεδρε, νομίζουμε ότι κλειδί για το μέλλον θα είναι η απασχόληση. Έχουμε μέχρι στιγμής ανεργία που φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ, κυρίως ε, στους νέους. Ε, κάτω των 25 οι νέοι έχουν αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας, ε, πάνω από 23% μερικές φορές. Όταν μιλούμε για οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να ξεχνούμε αυτή την κοινωνική ομάδα των νέων ανθρώπων γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε απασχόληση και για αυτούς. Ε, παρά και εξαιτία τη ύφεση υπάρχουν όλο και λιγότερε προσφορέ θέσεων εργασία. Ε, Δυστυχώ, άνθρωποι πτυχιούχοι ε, μένουν εκτό θέση εργασία, κάτι που αποτελεί τεράστια απώλεια και για την οικονομία μα. Έχουμε και άλλη ομάδα δανέων των ανειδίκευτων, χωρί ιδιαίτερα επαγγελματικά προσόντα. Και είναι δύσκολο στα κράτη-μέρη να ε, επενδύσουν στην παιδεία εξαιτία τη περικοπή των προπολογισμών. Εκεί μα έχουν οδηγήσει οι δημοσιονομικέ περικοπέ και η λιτότητα. Και μάλιστα η κατάσταση θα αυξηθεί ε, αν ε, με τις δημοσιονομικές προοπτικές υιοθετήσουμε το λιγότερο φιλόδοξο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σιμάνσκι. Επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Ινέ Κριστίνα Ζουμπέρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι μαγικές ρετσέτες της εξυγίανσης θα μπορέσουν να οδηγήσουν οικονομική ανάπτυξη. Η πραγματικότητα είναι στο πλαίσιο αυτό που βρισκόμαστε έχουμε δύο αντιθετικές απόψεις. Υπάρχουν οι οικονομολόγοι που λένε ότι χρειάζεται να υπάρξει δημόσια επένδυση και αύξηση της κατανάλωσης για να υπάρξει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δείχνει κάθε μέρα ότι υπάρχει μεγάλη δυσφορία, μεγάλα βάσανα που περνάνε οι οικογένειες στην Ευρώπη. Υπάρχουν οικογένειες που χάνουν την οικονομική επιδότηση από επιδόματα, από κοινωνικές παροχές. Χάνεται λοιπόν η κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν μπορεί μόνο η οικοδομία να το κάνει αυτό. Η Πορτογαλία βρίσκεται σε μια κατάσταση που έχει χάσει σχεδόν 10% του ΑΕΠ της. Όλο και περισσότερο χάνονται θέσει εργασία, 600 την ημέρα. Είναι απαραίτητο να αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Πρέπει να υπάρξει βιομηχανοποίηση, να ενισχύσουμε τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, να αυξήσουμε τους μισθούς και τις ε, συντάξεις και να ξαναγυρίσουμε τα κονδύλια από τον χρηματοπιστωτικό τομέα στους εργαζόμενους. Πρέπει επομένως να αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο τις νέες πολιτικές. Ζουμπέρ, καλώ βήμα τη συνάδελφο κυρία Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κυρία αντιπρόεδρε της ευρωπαϊκής επιτροπής συνάδελφοι ελπίζω ότι αυτά που συζητούμε σήμερα εδώ και τα μηνύματα που στέλνουν οι συνάδελφοι να είναι ενδιαφέροντα όχι μόνο για την ευρωπαϊκή επιτροπή αλλά και για το ευρωπαϊκό συμβούλιο που συνέρχεται σύντομα άμεσα στις ε, βρυξέλλες. Ε, το θέμα της ανάπτυξης δεν είναι βέβαια το θέμα του ευρωπαϊκού συμβουλίου αλλά δεν ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη είναι ο μεγάλος ασθενής βρίσκεται στα θεμέλια της προσπάθειάς μας για τη βιωσιμότητα του πολιτικού και του οικονομικού μας σχεδίου και παράλληλα η ανάπτυξη είναι ο μοχλός που μπορεί να κινητοποιήσει η ευρωπαϊκή ένωση για την ανάκαμψη της οικονομίας την ανάταξη της κοινωνίας που υποφέρει χάνει την πίστη της στην ευρωπαϊκή ένωση ιδιαίτερα στις χώρες που υφίστανται βαριές συνέπειες της ύφεσης και της λιτότητας όπως η χώρα μου η ελλάδα και η νέα γενιά χάνει την πίστη στο αύριο οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για την ε, ε, επόμενη χρονιά για την ανάπτυξη τόσο για την ένωση και ιδιαίτερα για την ευρωζώνη. Ε, η ευρωπαϊκή ένωση εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος ο σημαντικότερος στο σύγχρονο κόσμο αλλά βρίσκεται σε φθήνουσα πορεία. ήδη πρόσφατες ανακοινώσεις μας λένε ότι η κίνα το 2030 θα είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και φαίνεται το 2030 να μην είναι τόσο μακριά και φυσικά μέχρι να φτάσουμε εκεί θα έχουν προηγηθεί διάφορες ε, ανακατατάξεις ε, ε, στον κόσμο. αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε ότι η ευρωπαϊκή ένωση δεν κατάφερε να βρει την ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής εξυγίανσης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής είναι λοιπόν καιρός να δούμε πώς στις προτεραιότητες που έχει παρουσιάσει η ένωση για την επόμενη χρονιά θα μπορέσουμε να κάνουμε τις διορθωτικές παρεμβάσεις διότι δεν είναι δυνατόν να δικαιολογήσουμε τις αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των χωρών της ένωσης με όλες τις συνέπειες που έχουν για την προσπάθεια ανάκαμψης αποκλίσεις ως προς την ε, ε, ε, ε, πρόσβαση στη ρευστότητα αποκλήσεις ως προς την ζωντάνια της αγοράς εργασίας τα ποσοστά απασχόλησης είναι στοιχεία τα οποία δυναμητίζουν την προσπάθεια των χωρών που υφίστανται το βάρος της ανάκαμψης και παράλληλα την ίδια την ένωση γιατί χωρίς σύγκληση και συνοχή δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους της. ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ κυρία κράτσα. Κυρία Κράτσα, ο συνάδελφος κύριος Πάουλ Ρίμπιχ θέλει να κάνει χρήση της μπλε κάρτας. Αποδέχεστε το αίτημά του. Κύριε, κύριε Ρίμπιχ. Äh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή συζητούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, Ανάπτυξη και Απασχόληση. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα της Ευρώπης 2020 είναι ικανοποιητικό σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι θα πρέπει εκεί να τεθεί μια προτεραιότητα από το Συμβούλιο και επομένως ένα κατάλληλο ποσοστό του προϋπολογισμού να αφιερωθεί και σε αυτόν τον στόχο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντική ε, και θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό που υπονοείτε κύριε συνάδελφε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να τύχουν του κατάλληλου κλίματος τόσο από τις πολιτικές τις ευρωπαϊκές όσο και από τις εθνικές και όταν είπα στην παρέμβασή μου για την πρόσβαση και ε, την δυσκολία στην πρόσβαση στη ρευστότητα και κυρίως την ε, άνηση κατανομή στην ευρωπαϊκή ένωση σημαίνει ακριβώς ότι αυτό φύγει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. πρέπει να δούμε ότι είναι ο μοχλός αυτού του μοχλού που ανέφερα ότι χρειάζεται να κινητοποιήσει η ευρωπαϊκή ένωση για την ανάκαμψή της. Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος και έχει το Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Χουάν Γκόκ είπε ότι την Παρασκευή δημοσιεύθηκαν στους Financial Times ένα άρθρο το οποίο δείχνει πραγματικά τι σημαίνει ε, η Ισουητισμός. Αυτός που το έγραψε είναι ο Επίτροπος Αντιπρόεδρος Ρένα. Τι διαβάζαμε στα αγγλικά μια χώρα μπορεί να έχει περισσότερο χρόνο, να της δοθεί περισσότερος χρόνος για τα υπερβολικά ελλείμματα, για να τα διορθώσει. Ή μπορούμε επίσης να δεχθούμε και τις δημόσιες επενδύσεις στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας προβλέψεων ή επίσης ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τη δημοσιονομική εξυγίανση. Οπότε ο Αναγνώσης λέει ότι υπάρχει μια κίνηση εδώ, κάτι αλλάζει. Κάποιες έστω αμφιβολίες υπάρχουν για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής λιτότητας. Όχι βέβαια, στην κλασική ρητορική, δεν υπάρχει τίποτα το απροσδόκητο, λέει στα ελληνικά ο ομιλητής. Ε, στην ουσία περιμέναμε, είχαμε μία φιλοδοξία, μία προοπτική η οποία συστηματικά διαψεύδεται αλλά εμένουμε σε αυτή, λέει ο Πρόεδρος. Εμείς θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία. Αυτός επιμένει, όχι θα μείνουμε στην ίδια πορεία. Αυτό είναι πραγματικά η ισουητισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην ουσία έχουμε σε σύγκρουση ανάμεσα στον 18ο και το 19ο αιώνα, ανάμεσα στους γιανσενιστές, τους αυστηρούς, οι οποίοι πίστευαν ότι στο τέλος ο Ισουητισμός του Ρένερ θα μπορούσε να υποτιμήσει κατά κάποιο τρόπο ε, και να ελαχιστοποιήσει το αμάρτημα των χωρών οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι χρεωμένες. Ας επιλέξουμε λοιπόν τον τρίτο δρόμο. Κίνητρα, πολιτική με οικονομική δυναμική, ρεαλιστικούς επιτεύξιμους στόχους, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σωστή ρεαλιστική αντιμετώπιση του χρέους και του ελλείμματος. Πολύ κύριε Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Για Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε χαιρετίζω αυτή την ευκαιρία για να μιλήσω για την σημασία μιας συνολικής αντιμετώπισης στην ανάπτυξη. Τα μέτρα τα οποία προτείνονται από την Κομισιόν θα πρέπει όμως να συμβαδίζουν με τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση ανεργίας ιδίω των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν 22% το επίπεδο ανεργίας των νέων στην Ευρώπη με χώρες οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ και φτάνουν το 50% στη χώρα μου την Ιρλανδία ιδιαίτερα έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η ανεργία των νέων. 7,5 εκατομμύρια νέοι μεταξύ 18 και 29 δεν ήταν σε απασχόληση ούτε σε κατάρτιση ή εκπαίδευση. Για τα άτομα αυτά η προοπτική είναι ότι τα εισοδήματά τους δεν θα φτάσουν ποτέ τα επίπεδα που προσδοκούν. Αυτό θα οδηγήσει σε απογοήτευση και απόγνωση για πολλού. Είναι μια χαμένη γενιά για πάρα πολλού. Για να υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη, να υπάρξουν δράσει σε όλα τα επίπεδα για να αντιμετωπιστεί αυτό το αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, προτού να είναι μη αναστρέψιμα τα αποτελέσματα αυτή τη κατάσταση και οδηγήσουν σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτοί οι νέοι θα πρέπει να έχουν μια ευκαιρία να συμβάλλουν στην οικονομία και να μπορέσουν να αποκομίσουν τον σεβασμό των άλλων και να έχουν και μια δέσμευση εξ των λήπτων αποφάσεων. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να κάνει κάτι για αυτή τη γενιά. Μια τέτοια πρωτοβουλία χρειάζεται ηγετικό ρόλο και δέσμευση από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να έχει πραγματικό αποτέλεσμα και μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πρωτοβουλίε μα έναντι των νέων θα δώσουν πραγματικά αποτέλεσμα και θα είναι κενά λόγια μονάχα. Aylward, επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Μαρτίνα Άντερσον. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, δυστυχώς ε, εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στο κατόφυλλο της φτώχειας με όλο και επιδεινούμενες βιωτικές συνθήκες. Και μάλιστα το χρέος των τραπεζών ε, το υπομίστηκαν οι φορολογούμενοι που, σε χώρες που δυστυχώς ε, βρέθηκαν εκτός κεφαλαίου αγοράς. Ε, μέχρι στιγμής οι πολιτικές μας όχι μόνο δεν έλυσαν το πρόβλημα, αλλά το επιδίνωσαν. Και οι τράπεζες που έχουν ρευστό θα έπρεπε να υποχρεωθούν να δανείζουν για καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη για να βρεθεί το κεφάλαιο αυτό που χρειάζεται για να οδηγηθούμε στην ανάκαμψη και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Δεν οφείλεται κάτι τέτοιο σε έλλειψη δημοσιονομική ε, πειθαρχία. Δεν μπορούμε να έχουμε σωστό ισολογισμό με μαζική ενέργεια. Δεν μπορούμε έτσι να εξέλθουμε από την κρίση και να οδηγηθούμε σε οικονομική ανάπτυξη. Μόνο με πραγματικέ επενδύσει σε θέσει εργασία μπορούμε να επανέλθουμε στην πορεία τη ανάπτυξη και να μειώσουμε το δημόσιο χρέος ε, σε βιώσιμα επίπεδα. Ευχαριστώ. Αδελφός κυρία Μαρίτα Ουλσκοκ για λεπτό. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γνωρίζουμε όλοι και μάλιστα πολύ καλά πώς ξεκίνησε η κρίση. Από την έλλειψη ρύθμισης ε, στις κεφαλαίου ε, στην, ε, στις ΗΠΑ που τις αγάγαμε και στην Ευρώπη και μετά εφαρμόσαμε πολιτικές ε, που όξυναν την κρίση να την, την επιλύσουν. Υπάρχουν βέβαια τρόποι για να εξέλθουμε από το διέξοδο αυτό. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις κοινοτικέ αποφάσεις και να αξιοποιήσουμε το μέχρι στιγμή ανεκμετάλλευτο δυναμικό μας και μάλιστα για πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις ιδιαίτερα για επενδύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε και οικονομική ανάπτυξη και μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική για να αποφύγουμε ε, χειρότερες κρίσεις στο μέλλον. Το θέμα δεν είναι μόνο η πολιτική μας στόχη όταν μιλούμε για το κλίμα και το περιβάλλον. Είναι θέμα και πολιτικών και κοινωνικών στόχων. Με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων έχουμε δυστυχώς ε, ε, περικόψει τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους Κινέζους εργαζόμενους περικόπτοντας τους δικούς μας μισθούς. Δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στις περιβαλλοντικές μας προδιαγραφές. Θα πρέπει και οι υπόλοιποι να ακολουθήσουν το δικό μας δρόμο, γιατί εμείς έχουμε ειδικευμένου εργαζομένους που αξίζουν αξιοπρεπείς μισθούς. Γι' αυτό και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε κύριε συνάδελφε. Ακολουθεί στο βήμα η συνάδελφος κυρία Σίλβια Αντριάνα Τικάου. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Madam Commissioner. Κυρία Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κυρία... Τα θέματα που συζητούμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δυστυχώς, δυστυχώς, στο 2011 η ένδια και ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν αυξηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δραματικό τρόπο. Από 49% στη Βουλγαρία έχουν φτάσει το 49% στην Βουλγαρία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα ε, κίνηση επαναβιομηχάνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και επομένως να αυξήσουμε την κατάρτιση των νέων, κάτι το οποίο θα οδηγήσει και σε ένα νέο σύμφωνο ανάπτυξης. Μόνο λοιπόν με πολιτικές ε, λιτότητας δεν μπορούμε να προκαλέσουμε την οικονομική άνταξη. Εγώ χαιρετίζω την εισαγωγή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη ανάκαμψη για μη εκτό του τραπεζικού τομέα και έτσι θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ κυρία Τικάου, ανοίγει η διαδικασία Catch the Eye. Έχουν υποβληθεί δύο αιτήματα. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Πέτρο Λούχαν. într o perioadă în care problemele financiare persistă europa are nevoie mai mult eh, ca niciodată de măsuri urgente Έχουμε πολλέ δυσκολίε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, μεγάλη κρίση, γι' αυτό και κατεπηγόντω θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για να ανακτήσουμε την οικονομική μας ευημερία και να επανέλθουμε στη, στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις. Και ένα σημαντικό πρόβλημα που θα πρέπει να απασχολήσει κατά προτεραιότητα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κίνδυνο τη αποβιομηχανοποίηση τη Ευρώπη. Γιατί χωρί βιομηχανική βάση, χωρί ισχυρό βιομηχανικό ιστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει καμία δυνατότητα να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη έγιναν σημαντικές περικοπές στις βιομηχανικές επενδύσεις θα ε, έξω του 2,5% του ΑΕΠ. Θα πρέπει να ανακτήσουμε την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, να τις επαναφέρουμε στα εργοστάσια μας. Αλλιώς αποκλείεται να ανταγωνιστούμε τις βιομηχανικές υπερδυνάμεις. Θα συρρυκνωθεί η ανταγωνιστικότητά μας και ο ρόλος μας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Das Wort hat nun Herr Kollege Äh, äh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ΣΤΟΑ, ο φορέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις τεχνολογικές επιλογές, είχε την ευκαιρία και στο παρελθόν να βοηθήσει στο νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πράγματι ασχολήθηκε με το θέμα του ποιες είναι οι τεχνολογικές επιλογές επιλογές που χρειάζονται για μεγαλύτερη κινητικότητα, για, όπως είναι η πρωτοβουλία Connecting Europe, για μεγαλύτερη χρήση τη ψηφιοποίηση. Επίση και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας θα πρέπει και αυτό να εξασφαλίσει τη μεταλαμβάνευση των γνώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξει μεγαλύτερη γνώση και χρησιμοποίηση τη γνώση στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία ώστε με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε μαζί με την κινητικότητα και την κινητοποίηση των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσουμε την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας από την εκκίνηση μέχρι τον τελικό καταναλωτή και με τον τρόπο αυτό να δημιουργήσουμε περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη με την καλύτερη χρήση του διαδικτύου και έτσι επίσης να εξασφαλίσουμε και με την καλύτερη υγεία των πολιτών όπως το πρόγραμμα Perfect Life ότι θα συμβάλλουμε σε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε ε, Ρούμπιχ. Και τώρα ο κύριος Κονφράτη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να αναφέρω και μόνο προς την κυρία Επίτροπε ότι υπάρχουν δύο προβλήματα στην κατάσταση κρίσης την οποία διατρέχουμε έχουν αναφερθεί, αλλά νομίζω ότι θέλω να τονίσω το πόσο επικίνδυνα είναι. Επειδή δεν υπάρχει αρκετή απασχόληση, πολλές φορές μιλάμε για το πρόβλημα της απασχόλησης και αναφέρουμε τη μείωση της απασχόλησης σαν κύριο σύμπτωμα και πρόβλημα. Ξεχνάμε όμως την αύξηση της ένδυας. Η ένδυα γίνεται μια κατάσταση πραγματικά έκτακτης ανάγκης σε πάρα πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τόσο επικίνδυνη η ένδυα γιατί συνδέεται και με μια εξέλιξη που είδαμε στι ΗΠΑ αλλά που έρχεται και στην Ευρώπη. Είναι η πτωχοεργασία, όπω λέμε. Υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εργάζονται και δεν καταφέρουν με τα εισοδήματα από την εργασία να ξεπεράσουν το κατόφλι τη ένδυα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ω το κύριο πρόβλημα, γιατί έχει πάρα πολύ σημαντικέ επιπτώσει σε ό,τι αφορά την έλλειψη απασχόληση. Θα πρέπει να αποδοθεί λοιπόν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα και να θεσπιστούν οι κατάλληλε πολιτικέ. είναι ο κύριος Μασίπ. απέναντι σε τόσο παράλογη λιτότητα και τώρα που μιλούμε για τις απαρχές της Ευρώπης θα πρέπει να σκεφτούμε και τις δικές μας ρίζες γιατί η Ευρώπη σφυριλατήθηκε με την πρόσπιση του άνθρακα και του χάλιβα. Θα πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν στην προστασία της βιομηχανίας του άνθρακα και της χαλιβουργίας και να μην επιτρέψουμε τη μετακατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίστε περιομένη η συζήτηση. Διακόπτουμε ως την 12η μεσημβρινή ώρα των ε, ψηφοφοριών. Ε, δεχτείτε σας παρακαλώ τις ευχές μου για καλά Χριστούγεννα και ευτυχές στο νέο έτος. Merry Christmas and Happy New Year.